Αγαπητοί συναδελφοί, συνεχίζουμε. Τώρα η μερίστη διάταξη προβλέπει δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σχετικά με ξένε επενδύσει σε στρατηγικού τομεί. Το λόγο έχει η κυρία Ντάλη, εκ μέρου του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη δεδομένου ότι το θέμα των ξένων επενδύσεων σε στρατηγική τομή είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί αυτό καθ' αυτό στο Συμβούλιο ακόμα. Συνεπώς δεν υπάρχει θέση του Συμβουλίου ακόμα.